Oh. Angelis on the Schademoser report. Mr. De Angelis. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σάρλμος ε, για την έκθεσή της ε, που κατά κύριο λόγο έχει ως στόχο να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων εποπτείας, κυρίως όσον αφορά την διακίνηση στην ευρωπαϊκή αγορά ασφαλών προϊόντων για τους Ευρωπαίου καταναλωτές. Είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και αφορά στην ολοκλήρωση της κοινή αγοράς και στην προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών. Τον διασφαλίζει κανείς την ασφάλεια σημαίνει ότι πρέπει να έχει μηχανισμούς ίχνηλασιμότητας, να παρακολουθεί όλη τη διάρκεια, όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Άρα δηλαδή αποτελεσματικές προτάσεις, δημιουργία ε, τράπεζα δεδομένων για την ασφάλεια των προϊόντων, προϊόντων, ενίσχυση του συστήματος RAPEX κυρίως όσον αφορά τα επικίνδυνα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες ε, χώρες. Ε, να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές εποπτείας να διασφαλίζουν στην αγορά προϊόντα χωρίς κινδύνους. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι η δική μας η δουλειά είναι να εγγυόμεθα ότι τα προϊόντα που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή αγορά ε, να είναι ασφαλή για τις ευαίσθητες κατηγορίες ανθρώπων όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι ανάπηροι. Κύριος Καλινόφσκι. Ευχαριστώ. Πολλά λέμε για την ασφάλεια των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, αλλά μερικές φορές ξεχνάμε και τα προϊόντα καθημερινής χρήσης που πολλές φορές περιέχουν κινδύνους σοβαρές και σοβαρές απειλές για τη ζωή, ιδιαίτερα των παιδιών. Και μάλιστα είναι μεγάλη πρόκληση με τα προϊόντα εισαγωγής. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος και μάλιστα εποπτεία και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Με συνεργασία των οργανώσεων προστασίας καταναλωτών και των εθνικών αρχών θα προχωρήσουμε, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και τον ορισμό του ασφαλούς προϊόντος, χωρίς να ξεχνάμε και το σωστό σχεδιασμό των οδηγιών χρήση, αλλά και το σύστημα ασφάλεια των διαφόρων προϊόντων. Και φυσικά θα πρέπει να έχουμε υπόψη την λογική χρήση του, αλλά και να έχουμε υπόψη και την ασφάλεια των παιδιών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κόμη. Κυρία Πρόεδρε, σήμερα το Κοινοβούλιο ψήφισε για το θέμα τη ασφάλεια των προϊόντων. Ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αποτελεί ένα βήμα προ τα εμπρό που αφορά στην ενίσχυση τη προστασία του Ευρωπαίου καταναλωτή. Οι εκθέσει που έγιναν υπογραμμίζουν τη σημασία τη συχνηλασιμότητα για όλο τον κύκλο ζωή των προϊόντων και καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, παρακολουθεί την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Ε, πρέπει λοιπόν ε, να βελτιστοποιηθεί και το κόστο προ όφελο του καταναλωτή. Ο Ευρωπαίος καταναλωτής έχει το δικαίωμα να γνωρίζει όλα τα στοιχεία του προϊόντος γιατί με τον τρόπο αυτό αισθάνεται περισσότερο προστατευμένος. Πιστεύω λοιπόν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στον αγώνα κατά της παραποίηση ε, κυρίως στον, ε, στον τομέα της κλωστεφαντουργίας. Πρόκειται για την προστασία του καταναλωτή αλλά και όλων εκείνων των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ευρώπη και που δεν έχουν αποφασίσει να αναθέσουν σε τρίτους τις δραστηριότητές τους. Θεωρώ ότι μπορούμε λοιπόν να βρούμε μια βέλτιστη λύση όσον αφορά κυρίως ε, την ονομασία των προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρε, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη ιχνηλασιμότητα. Για την επόμενη έκθεση ε, για την διαχείριση της γρήπης, ο κύριος Μπαρτελότσι. Κυρία Πρόεδρε, ε, υπέρ υπερψήφισα γιατί θεωρώ ότι πράγματι πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση της γρήπης ή τα ή ε, μία διαχείριση που θα έχει ως στόχος ε, να υπάρχει ε, καλύτερη συμπεριφορά κυρίως σε σχέση με το ενδεχόμενο να υπάρξουν στο μέλλον έκτακτες καταστάσεις. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει συνεργασία, ανεξαρτησία και διαφάνεια. Αυτές είναι οι βασικές αρχές και όλα αυτά έχουν ως στόχο την καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε πραγματικά να μην υπάρξει κίνδυνος και να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση. Η στόχη είναι να εναρμονιστεί η στρατηγική των κρατών μελών κυρίως αναφορά τα προγράμματα εθνικής διαχείρισης την ε, δημοσίευση των απαραίτητων στοιχείων. Ε, πρόκειται για μια σχέση εμπιστοσύνη με τα μέσα ενημέρωση τα οποία έχουν ως στόχο να μεταφέρουν τα μηνύματα για τα θέματα και γι' αυτό εγώ υπερψήφισα. Κυρία Μάτιες. Ευχαριστώ. Γνωρίζουμε τι συνέβη με την γρήπη Α και θα έπρεπε να μας γίνει το πάθημα μάθημα. Δεν ξέρω αν θυμάστε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ξεκίνησε με έναν τρόπο, αλλά η απάντηση ήταν τελείως δυσανάλογη σε σχέση με τις διαστάσεις του προβλήματος. Γι' αυτό και η σημερινή έκθεση Ριβάζη είναι πολύ σημαντική, γιατί θα πρέπει να μάθουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος και να μην επαναλάβουμε τα προηγούμενα λάθη. Θα πρέπει να δούμε πώς έλειψαν οι αποφάσεις, πώς συνέβησαν όλα αυτά και τι ήταν αποφασιστικό για να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Ορισμένες χώρες ανταποκρίθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί όμως διάλεξαν αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτή η αδιαφάνεια. Γιατί παρά τις αφιβολίες που εκφράσαμε δεν διασκεδάστηκαν. Νομίζω ότι θα πρέπει να διελευκανθεί η κατάσταση σε σχέση με την γρήπη και φυσικά να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της υγείας, αλλά ο τρόπος είναι πολύ σημαντικός, γιατί έχει και κάθε τρόπος έχει συγκεκριμένο τίμημα. Ο κύριος Γκζίμπ. Ευχαριστώ. Η έλλειψη ανεξάρτησης αξιολόγησης από τα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι το θέμα και μέρη της έκθεσης Ριβάση ε, για τη διαχείριση της γρήπης ΙΤΑ 1 1 1. Μερικές φορές ε, γίνονται, λαμβάνονται ακατάλληλες αποφάσεις ε, για θέματα υγείας. Και μάλιστα ακούσαμε από ηθινόντα ότι πότε προηγουμένως δεν είχαμε τέτοια ε, μαζική χρήση εμβολίων και μαζικό εμβολιασμό σε παρόμοια ζητήματα στο παρελθόντα. Επίσης, τι γίνεται ε, και με, την, ε, με τα διάφορα στοιχεία του, εμβολίου. Ήταν αδιαφανή η διαδικασία λύση αποφάσεων παρά το πολύ σημαντικό θέμα στην Πολωνία. Η Υπουργό Υγεία υπέστη πιέσει και από τα μέσα μαζική ενημέρωση και τελικά δεν έλαβε την απόφαση για την αγορά των εμβολίων και για το μαζικό εμβολιασμό. Επίσης, ε, καθημερινά πανικοβάλλονταν οι πολίτες εξαιτία του βομβαρδισμού που πέσαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ανάγκη εμβολιασμού. Θα πρέπει να δούμε τα υπέρ και τα κατά, γιατί το κέρδος δεν είναι το σημαντικότερο. Η ασφάλεια των καταναλωτών και των ασθενών είναι το σημαντικότερο. Γιατί τα εμβόλια όντως θα πρέπει να μας αποτρέψουν και να μας γλιτώσουν από τις ε, ε, από τα προβλήματα υγείας. Έχουμε πάνω από 50 επεξηγήσεις, ε, αλλά και εγώ πεινάω και οι διερμηνείς μας δικαιούνται το γεύμα τους. Παρακαλώ μην ξεπερνάτε το χρόνο αγόρευσης, γιατί είχαμε μια παρατεταμένη ψηφοφορία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε και το χρόνο αγόρευσης. Κύριε Σαντινόρη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μέχρι σήμερα η σύσταση που έχει εγκριθεί ε, για τα ε, ετναλία την στη Μεσόγειο ε, αφορά τις αιτήσιες ποσοστώσεις. Εδώ λοιπόν πρόκειται για την διαχείριση, τον έλεγχο, την ε, εμπορία των προϊόντων αλίας στη Μεσόγειο. Ο μόνιμος ε, χαρακτήρας ε, της σύστασης απαιτεί βέβαια να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα, κυρίως όσον αφορά το κοινωνικό δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει μια ενιαία νομοθετική πράξη όπου θα αναφέρονται όλες οι μελλοντικές συστάσεις. Σήμερα λοιπόν κάναμε ακριβώς αυτό και με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί το δίκαιο το οποίο ε, σίγουρα θα οδηγήσει σε απλουστεύσεις. Τα συμβαλόμενα μέρη της CGMPM έχουν το καθήκον να διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή ε, των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί και επίσης ε, και την έγκυρη μεταφορά του σε εντρικό δίκαιο έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να ισχύουν για νομικά και φυσικά πρόσωπα σε κοινοτικό, σε κοινοτικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Η ομάδα μας υποστήριξε την έκθεση αυτή, γιατί είναι πολύ σημαντική στα πλαίσια του σχεδιασμού και της εφαρμογής της μελλοντικής κοινωνικής κοινοτικής ελευτικής πολιτικής. Το θέμα της περιφερειοποίησης είναι πολύ σημαντικό και η στήριξη της ΚΑΠ στην ε, περιφερειοποίηση και την αποκέντρωση είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει και το θέμα των απορρίψεων βέβαια, ε, δεν θα πρέπει να το παραλείψουμε από τη συζήτηση ιδιαίτερα στα πλαίσια της περιφερειοποίησης και της αποκέντρωσης. Γι' αυτό και με αυτές τις βάσεις θα πρέπει να χτίσουμε την κοινή αλληλευτική μας πολιτική. Ευχαριστώ κύριο Κεμάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν κοιτάξουμε την ιστορία το ιστορικό στην κοινή γεωργική πολιτική αλληλευτική και τις διεθνείς συμφωνίες, το αποτέλεσμα είναι σαφές. Ε, ορισμένες περιοχές εξωθούνται στην αύξηση της παραγωγής με τεχνητές τιμές το ίδιο ε, το πρόβλημα έχουμε και με τα αποθέματα των αλλιευμάτων. Με τις απορρίψεις ε, έχει αποτύχει αυτό το σύστημα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχουν δικαιώματα τα οποία να μεταβιβάζονται και, για να εξασφαλίσουμε και τις σημερινές γενναίες και τις περχόμενες. Αν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε το κράτος δικαίου, τα κυριαρχικά δικαιώματα και στις αλλίες, θα έχουμε η πολιτική όχι μόνο για την αλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παγκόσμια και δεν θα χρειαζόμαστε καθόλου τέτοιες συμφωνίες. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Κάθε μέρα ε, χιλιάδες ε, ε, τόνοι νεκρών ψαριών απορρίπτονται στη θάλασσα από τα σκάφη. Και ε, ως ε, πτώματα ψαριών πέφτουν ε, και βυθίζονται στη θάλασσα και ρηπαίνουν και το βυθό. Και είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό των απορρίψεων. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσει. Το κατάλαβε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά οποιαδήποτε λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, έχει προβλήματα. Ε, μπορείτε να περιορίσετε το μάτι, το μέγεθος των δικτύων, μπορείτε να περιορίσετε τις ημέρες αλίευσης, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά όλα αυτά βασίζονται στο υπαρξιακό πρόβλημα, στο λόγο ύπαρξης της κοινής αλλιευτικής πολιτικής, ότι είναι κοινή αυτή η πολιτική, ότι θεωρείται ότι είναι ένα κοινό αγαθό και κανένας δεν το αισθάνεται κτήμα του και κανένας δεν έχει την ε, πρωτοβουλία ή το κίνητρο να το κοιτάει ε, ως ένα ε, είδος που θα πρέπει να διαφυλάσσεται και να ανανεώνεται. Αυτό θα γίνει μόνο με εθνικούς, εθνική κυριαρχία στα χωρικά μας ύδατα. Ε, ο κύριος Ρόντε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών στο Κοινοβούλιο και πάλι θεωρεί ότι θα πρέπει εμείς να, να επιβάλλουμε ένα νέο φόρο τώρα στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Αυτός ο λεγόμενος φόρος Τόμπιν από όλους τους φόρους που γνωρίζουμε είναι ο πιο ηλίθιος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν πρόκειται να επιβληθεί. Διότι αλλιώς θα είχε επιβληθεί εδώ και καιρό γιατί όπως γνωρίζετε για πρώτη φορά προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 ήδη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ε, ξανά έγινε αυτή η πρόταση και μετά από λίγο χρόνο θα έρθουμε να διαπιστώσουμε ότι δεν ήταν και τόσο καλή σκέψη και δεν είναι καλή ιδέα όντως ε, να επιβάλλουμε στην Ευρώπη ένα τέτοιο τέλος ή ένα τέτοιο φόρο διότι τα χρήματα μπορούμε να τα ε, ε, βρούμε από αλλού στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτός ο φόρος Τόμπιν δεν είναι η λύση για οτιδήποτε στην Ευρώπη. Αυτό το κατάλαβε και ο ίδιος ο Τόμπιν και το αναγνώρισε πριν από λίγα χρόνια. Presidente, Κύριε Πρόεδρε, η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει αποδείξει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις όσον αφορά τις ρυθμίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομική κρίση ήταν μια πολύ ευαίσθητη κρίση προπολογισμών και κρίθη απαραίτητο να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα για να μπορούν τα κρατημέλη να εκπληρώσουν ε, τις υποχρεώσεις τους. Ε, για άλλη μια φορά λοιπόν ελήφθησαν βραχυπρόθεσμα μέτρα ε, στο επίκεντρο της Κρήτης και αποδείχτηκε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στην εποπτεία και τα δημόσια οικονομικά η κόστο αυτή τη κρίση δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί πλήρω. Εν πάση περιπτώσει έχει καταστεί απολύτω σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και γενικότερα ο κόσμο δεν μπορούν να επιτρέψουν άλλη μια κρίση και δεν μπορούν να επιτρέψουν να υπάρχουν τέτοιου είδου φαινόμενα. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε καινοτόμα στοιχεία, καινοτόμου μηχανισμού για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε και να αλλάξουμε και με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω την ε, επιβολή ενός τέτοιου παγκοσμίου όμως τέλους στις οικονομικές συναλλαγές. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει πρώτα μια εκτίμηση, μια μελέτη, ένα τέτοιο φόρος μπορεί να επιβληθεί σε πρώτη φάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από εκεί και πέρα με βάση αυτή τη μελέτη να λάβει απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Λονδίνο έχουν επιβάλει φόρο στο χρηματιστήριο και εισπράττουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Πολύ περισσότερα από αυτά που θα εισπράττουμε εμείς από το συγκεκριμένο τέλος. Και είναι θερεντικά λοιπόν τα όσα συμβαίνουν στο Λονδίνο και θετικά και χαίρομαι και θα το δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ γρήγορα να κάνει τέτοια μελέτη. Για ένα λεπτό. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, η οικονομική κρίση η οποία τα τελευταία χρόνια έπληξε την Ευρώπη, η κρίση αυτή επέδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε νέα εργαλεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε φρένο στην κερδοσκοπία και να επαναφέρουμε το ρόλο του χρηματοψητικού τομέα. Οφείλουμε να γνωρίζουμε πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες τη πραγματικής οικονομίας και να στηρίξουμε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό να υπάρχει και μια κατανομένες επιμερισμός ε, ε, του βάρους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να επιτύχουμε επιπρόσθετους πόρους για να αντιμετωπίσουμε τις ε, παγκόσμιες προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή αλλά και άλλα θέματα που έχουν αναφερθεί και αναφέρονται στη στρατηγική του 2020. Εγώ λοιπόν εύχομαι να αποδοθεί μεγαλύτερη σημασία στα μέτρα δημόσιου ελέγχου και στη διαφάνεια των καινοτόμων εργαλείων. Γιατί τα τελευταία κυρίως είναι μια συνεκουανόν προϋπόθεση για να μπορέσουμε μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ένα λεπτό. Signor Presidente, Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η έγκριση της ε, έκθεσης ε, της κυρίας Ποδηματά είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός ε, για μια οικονομική, φορολογική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μεγαλύτερη ισορροπία και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Είναι σαφές για όλους ότι είναι απαραίτητο ως Ευρώπη να επιτύχουμε ένα συντονισμό ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη, να καταλήξουμε στα απαραίτητα τα οικονομικά μέσα έτσι ώστε να ε, διαχειριζόμαστε την οικονομία και όχι απλά να την υφιστάμετα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι σωστά έλαβε χώρα όλη αυτή η συζήτηση σχετικά με την πρόταση περί ε, του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ενέκρινε αυτόν τον κανονισμό είναι ένα σημαντικό στοιχείο γιατί για πρώτη φορά δεν αφήσαμε να συμπαρασυρθούν Ευχαριστούμε. Κάναμε ένα βήμα προ τα εμπρό και εύχομαι η Επιτροπή του Συμβούλου να ακολουθήσει αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Μάριο, κύριο Σπυρίλο, για ένα λεπτό. Signor Presidente, grazie. L'attuale crisi Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η οικονομική κρίση κατέδειξε τις ε, ελλείψεις του συστήματος ελέγχου του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η αναγκαιότητα να αντιδράσουμε με νέα εργαλεία και νέες πολιτικές ε, κατέστη απόλυτα σαφής. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα άρχισε να ε, αποφέρει κέρδη από κερδοσκοπίες και είναι λοιπόν παράλογο ο τομέας αυτός να μην υφίσταται κανένα έλεγχο. Είναι απαραίτητο να υπάρχει θεραπεία και ένας φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Γι' αυτό λοιπόν εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Για πολιτικές όπως αυτή της ενέργειας και του περιβάλλοντος η Ευρώπη προηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο και δίνει το παράδειγμα ε, αυτό αποτελεί κίνητρο και για άλλα κράτη εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να γίνει και με τον χρηματοψηφιακό τομέα. Εύχομαι λοιπόν η Κομισιόν να αντιδράσει σύντομα και να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση έτσι ώστε να καλύψει τι ανάγκε ε, των ε, πολιτών, του οποίου έχει πλήξει κρίση. Για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η εφαρμογή ενό ε, νέου ε, φόρου, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε πολύ. Από τη μια, ε, επιτρέπει βέβαια να υπάρξουν κίνητρα και έτσι να περιορίζονται οι κίνδυνοι. Από την άλλη, όμω, δημιουργούνται στρεβλώσει που θα μπορούσαν να τιμωρήσουν τι οικονομικέ αγορέ στην Ευρώπη. Οι κερδοσκοπίε βέβαια θα πρέπει να φορολογούνται, αυτό είναι σωστό και θεωρώ ότι είναι σωστό να εξετάσει κανεί τα υπέρ και τα κατά. Γιατί ένα σε τέτοιος φόρος δεν είναι σωστά μελετημένος έτσι ώστε να αποδώσει τα ευκταία αποτελέσματα χωρίς όμως να τιμωρεί τους υπόλοιπους. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι σύμφωνα με τη λογική ότι αν η Ευρώπη λειτουργήσει και αντιδράσει μόνο θα χάσει ανταγωνιστικότητα και δεν θα έχει κανένα εργαλείο έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους άλλους παγκόσμιους παίκτες. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει φορολόγηση αλλά αυτή η φορολόγηση να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο κέρδισε ε, στους κόλπους της G20. Ε, Πρόεδρε, σήμερα εγκρίναμε με μεγάλη μας ικανοποίηση ε, την έκθεση της ε, κυρίας ε, Πόντιματα. Για μας λοιπόν, για την Ιταλική αντιπροσωπεία, την Ιτάλια Βαλόρι, για τη δική μας την πολιτική ομάδα, ήταν μια ιδιαίτερη ικανοποίηση. Γιατί το Κοινοβούλιο απέδειξε ότι ανταποκρίνεται σε θέματα αρχής. Υπήρξε μια συζήτηση για την έκθεση της κυρίας Μπερές για την κοινωνικονομική κρίση και τότε εμείς εκφραστήκαμε υπέρ του να υπάρχει ένα ένας ε, φόρος για τις ε, χρηματοψηφιακές συναλλαγές. Εμείς λοιπόν υπερψηφίσαμε αυτή την έκθεση της κυρίας Ποντήματα γιατί πρόκειται για ένα φόρο που θα βοηθήσει ε, να περάσουμε από την οικονομική κερδοσκοπία στην πραγματική οικονομία. Αυτή η έκθεση θα μας δώσει τη δυνατότητα, μάλλον τα μέτρα που θα ληφθούν θα δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουμε τους στόχους του 2020, να συμπεριφερθούμε με μεγαλύτερη φιλικότητα προς το περιβάλλον και να βοηθήσουμε με την παραγωγή. Περνάμε μια χρηματοπιστωτική κρίση και θα πρέπει να διδαχθούμε από τα παθήματά μας. Για παράδειγμα, η ε, ανεπαρκής νομοθεσία δημιουργεί προβλήματα. Ε, Στην Ηνωμένο Βασίλειο ε, ενθαρρύναμε τις τράπεζες να ε, χρηματοδοτούν ε, αφαιρέγγιους πολίτες. Έτσι όμως ξεκίνησε και η κρίση και είδαμε τις συνέπειες. Θα πρέπει να δούμε και τις συνέπειες της έκδοσης φθηνού χρήματος ή το ύψος των επιτοκίων, γιατί μερικές φορές ε, οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν την αξία του χρήματος και κάνουν κακές επενδύσεις. Ένας οικονομολόγος είπε με κακές αποφάσεις και κακές επενδύσεις θα βγούμε όλοι χαμένοι και θα έχουμε μια κρίση στην αγορά, αυτό που συνέβη. Δεν θα πρέπει οι τράπεζε ε, να έχουν την πολυτέλεια να αποτυχαίνουν επειδή λόγω του μεγάλου μεγέθους του και του οικονομικού τους βάρου. Γιατί αν δεν ε, μεριμνήσουμε θα συνεχίσουν ε, ασυλλόγιστα να δρούν οι τράπεζες. Θα πρέπει να διδαχθούμε από τα παθήματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. πρώτος ο κύριος Γιακολίνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σαφής απόδειξη ότι δεν είναι δεδομένο ακόμα το δικαίωμα στην ευρωπαϊκή ηθαγένεια ε, δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές στην υγεία στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει δικαίωμα ίσης περίθαλψης στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και δικαίωμα ουσιαστικό που να μπορεί κανείς να το επικαλείται. Είναι περίπλοκα τα ζητήματα και ε, σήμερα ε, εορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η πρόσβαση στην υγεία και την περίθαλψη είναι ακόμα πιο περίπλοκη για τις γυναίκες. Χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση, μεγαλύτερη πρόληψη ε, και καλύτερη ε, θεραπεία και καλύτερο στυλ ζωής. Μέθοδος, όχι στη στο αλκοόλ, όχι στην εξάρτηση, όχι στις ουσίες, όχι στην παχυσαρκία. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ως πραγματικό ευρωπαϊκό στόχο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάντα το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι η διατήρηση της υγείας και μετά η αποκατάσταση της υγείας και ενημέρωση σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή υγιεινή διατροφή και άσκηση. Αυτό είναι στοιχείο της βασικής εκπαίδευσης των γενικών γνώσεων και είναι υπόθεση των κρατών μελών. Η Ευρώπη θα πρέπει να προωθεί στην ανταλλαγή εμπειριών ε, για την περίθαλψη και για την ενημέρωση και την εκπαίδευση για την υγεία. Εγώ παρόλες αυτές τις καλές προθέσεις όμως καταψήφισα την έκθεση λόγω των παραγράφων 25, 26 και 29 γιατί εδώ οι σημαντικές αποφάσεις ηθικές και δεοντολογίας για την τεχνολογία αναπαραγωγής και τη διακοπή της κοίησης. Αυτό δεν έχει καμιά θέση εδώ μέσα. Είναι θέμα ε, των κρατών μελών και τα θέματα ε, της πρόληψης, προφύλαξης τα ζητούν ε, ξεκομμένα από το δικαίωμα στη ζωή. Arvoisa puhemies. Okay. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Στάκουλα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διαφορές και ανισότητες ως προς την προσέγγιση του θέματος υγείας μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν και διαφορετικές παραδόσεις και πρακτικές στην υγεία στα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε λοιπόν να γεφυρώσουμε αυτές τις ανισότητες και να περιορίσουμε τις διαφορές στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη κατάρτιση και επίγνωση του γεγονότος ότι αυτό που επηρεάζει την υγεία είναι και οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, όπως αναλύονται στην έκθεση. Πιστεύω πάντως ότι ε, η επικέντρωση μόνο στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην καλύτερη διατροφή, στον τρόπο άσκηση, αυτοί είναι πιο σημαντικοί παράγοντες και αυτού θα πρέπει να υπογραμμίσουμε αν πραγματικά θέλουμε μια υγιέστερη και καλύτερη Ευρώπη και να προβούμε και σε ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Εγώ δεν ψήφισα στην έκθεση αυτή γιατί ε, πιστεύω ότι περιλαμβάνει κάποια θέματα που είναι άσχετα με το περιεχόμενό της. Εμείς θα πρέπει να περιοριστούμε στο, στο γεφύρωμα αυτών των ε, διαφορών στο θέμα της υγείας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια μία από τις βασικότερες ανησυχίες μου όταν συζητούσαμε τη φορολογία σε διεθνές επίπεδο είναι επιθέσεις κατά των νησιών Καϊμάν για παράδειγμα ε, που το μόνο που έκαναν είναι να χρησιμοποιήσουν τις δικές μας συμβουλές για αναπτυξιακά θέματα. Λέμε στα νησιά της Καραϊβικής και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τις καλλιέργειές τους από τη ζάχαρη και τις μπανάνες και να ζητήσουν εμπειρογνωμοσύνη για θέματα υπηρεσιών. Αυτό έκαναν οι νήσοι Καϊμάν και τώρα 40 με 50% των υπηρεσιών τους είναι χρηματοπιστωτικέ χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες χάρη στο σύστημα φορολογικής ουδετερότητα, όχι φοροαποφυγής αλλά φορολογική ουδετερότητας. Δεν και τριπλασιάζουν τη φορολογία των ε, κονδυλίων που επενδύζουν εκεί. Οι υποκριτικοί περιληστές όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που αποφασίζουν είναι να ε, επιτίθεται στα νησιά Καϊμάν επειδή τολμούν ε, να ανταγωνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι τροπή αυτό για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ δύσκολο βρήκα να υποστηρίξω την έκθεση της φίλης κυρία Ζολή, διότι άρχισε να μιλάει για ένα φόρο ευρωπαϊκό στην αρχή και μετά παγκόσμιο. 818 δισεκατομμύρια δολάρια πηγαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες με διάφορους τρόπους νόμιμους και παράνομους και φεύγουν από τις χώρες αυτές και είναι καταθέσεις σε ευρωπαϊκές και δυτικές τράπεζες. Εμείς αντίθετα ε, ε, παίρνουμε χρήματα φορολογουμένων 60 με 70 δις και τα πηγαίνουμε ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες για να απαλληλθεί η φτώχεια. Αυτά τα 818 δισεκατομμύρια που φεύγουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες και είναι καταθέσει στις δικές μας τράπεζες, αν είχαν μείνει στις χώρες τους για να αναπτυχθούν οι χώρες αυτές, πόσο καλύτερα δεν θα ήταν τα πράγματα. Πιο γρήγορα αναπτυγμένοι θα ήταν και δικαιώματα θα είχαν και εμπορικούς φόρους. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση Παπαστάμκου. Πρώτος ο κύριος Μαστέλα για ένα λεπτό. Σε μια στιγμή κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να μεταρρυθμίσει την κοινή τη γεωργική πολιτική, να εγγυάται τη συνέπεια ανάμεσα στην γεωργική πολιτική και το εξωτερικό εμπόριο, ε, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη. Ε, Έχουμε λοιπόν ε, δύο πολιτικές ε, και η δυναμική τους γίνεται όλο και μεγαλύτερη, ασκούν όλο και μεγαλύτερη επιρροή σε παγκόσμιο, ε, σε διεθνές, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν μέσα σε διαπραγματεύσεις για να υπάρξει συμβασμός ανάμεσα στα εμπορικά συμφέροντα και το περίπλοκο της γεωργικής πολιτικής. Η γεωργική πολιτική δεν είναι μόνο οικονομική δραστηριότητα, αλλά είναι μια πολιτική η οποία έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις βασικές προκλήσεις ε, του σήμερα. Ε, έτσι λοιπόν η γεωργική πολιτική μπορεί να παίξει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να επιδιώκουμε τους στόχους μας ε, χωρίς να, υπάρχει, να θετεθεί σε κίνδυνος η δυναμική. Ευχαριστώ. η προτεραιότητα της κοινή γεωρικής πολιτικής είναι η ασφάλεια των τροφίμων. Για να γίνει εφικτή όμως η ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να υπάρχουν αναλογίες και έλεγχος του διεθνούς εμπορίου. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στον θεμητό και το δίκαιο ανταγωνισμό, γιατί οι, οι Ευρωπαίοι γεωργοί θα, ε, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν αυστηρές προδιαγραφές ε, και πολύ αυστηρούς κανόνες. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασκεί κανέναν απολύτως έλεγχο σχεδόν στους ε, γεωργούς και παραγωγούς τρίτων χωρών από τους οποίους εισάγουμε τεράστιες ποσότητες τροφίμων. Τέτοιου είδου εμπορικέ συμφωνίε είναι άδικε απέναντι στην τόπια παραγωγή, στην ευρωπαϊκή παραγωγή και μια τέτοια πολιτική είναι επικίνδυνη και για την υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών γιατί δεν έχουμε ουσιαστικό έλεγχο στην ποιότητα αυτών των προϊόντων. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι υπερψήφισα την έκθεση αυτή διότι πιστεύω ότι ε, αναφέρει πολύ καλά τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και των Ευρωπαίων αγροτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική. Η γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να θυσιαστεί για να κάνουμε ε, εμπορικές συμφωνίες ε, με τη Μερκοσούρα, ας πούμε. Ε, και δεν μου αρέσει αυτή η κατεύθυνση που παίρνουμε. Φαίνεται ότι υπάρχει αντίληψη ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό ε, ατού, ως μάρκα στην ε, οποία ποντάρουμε σε κάποια θέματα, ειδικά στην κτηνοτροφία. Σε ό,τι αφορά τις ίδιες προδιαγραφές, τις αντίστοιχες, ζητούμε να έχουμε τις ίδιες προδιαγραφές και για τις εισαγωγές, τα ίδια που απαιτούμε από τους παραγωγούς μας. Σίγουρα έχουμε ευθύνη απέναντι στους καταναλωτές να το διασφαλίσουμε αυτό. Και επίσης έμεινα πολύ δυσαρεστημένος από τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στο Κοινοβούλιο. Και ε, να ληφθεί υπόψη η άποψη Επιτροπής Γεωργίας. Είναι για ένα λεπτό. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος ε, Γκζιμπ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η έκθεση Παπαστάνκου καταλήγει σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές πολυμερείς και διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με το Παγκόσμιο Οργάνωση Εμπορίου και άλλες εμπορικές οργανώσεις. Ε, το εμπόριο έχει σημαντικό ρόλο για την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και μάλιστα είμαστε καθαρός εισαγωγέας ε, γεωρικών προϊόντων και ε, για τη ζάχαρη μετά την τελευταία ε, παραγωγή. Ε, αντί να είμαστε εξαγωγής όπως παλιά, γίναμε πλέον καθαρή εισαγωγή. Έχουμε 60% εισαγωγές γεωργικών προϊόντων. Έχουμε εμπορικό έλλειμμα σχέση με τη Λατινική Αμερική. Και μάλιστα εισάγουμε προϊόντα γεωργικά που στηρίζονται σε άλλες προδιαγραφές, πολύ πιο χαλαρές από αυτές που επιβάλλουμε στους ντόπιου παραγωγούς που πληρώνουν το βαρύ τίμημα της συμμόρφωσης με αυστηρή νομοθεσία. Η γεωρική πολιτική χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προπολογισμό. Δεν θα πρέπει όμω να μειώσουμε την αποτελεσματικότητά τη. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνέργεια μεταξύ τη κοινοτική γεωρική πολιτική και τη εμπορική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω λίγα λόγια για την έκθεση Παπαστάμκου. Είναι μια περιεκτική έκθεση και δίνει μια καλή εικόνα και κάνει μια καλή επισκόπηση για τον τρόπο λειτουργίας και συνέργειας μεταξύ της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής και της ε, εμπορικής πολιτικής. Μερικές φορές η γεωργία χρησιμοποιήθηκε για την άσκηση πολιτικής. Η γεωργία είναι σημαντικός κλάδος τη ευρωπαϊκή οικονομία και φυσικά όταν μιλούμε για κοινοτικέ πολιτικέ, η γεωργία βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Δεν θα πρέπει όμω να ξεχνούμε στο πλαίσιο αυτό ότι όταν ε, εισαγάγουμε τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να τηρούνται και κάποιε δεντολογικέ προδιαγραφέ. Για παράδειγμα, ε, η υγιεινή των προϊόντων είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η γεωργική παραγωγή στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο πληρεί πολύ αυστηρέ προδιαγραφέ. Στην ε, Φιλανδία παράγουμε καθαρά προϊόντα. Αυτή η σημαντική διοντολογική αρχή θα πρέπει να πρετανεύει και στην εμπορική πολιτική, όχι μόνο στη γεωργική. Ευχαριστώ. Εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης Παπαστάμκου και την εκτιμώ ιδιαίτερω ε, το περιεχόμενό τη Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ τη ασφάλειας ε, των τροφίμων ε, στην Ευρώπη και δυστυχώ, μερικέ φορέ αυτή η ασφάλεια των τροφίμων απειλείται από το Διεθνέ εμπόριο. Υπάρχει ισχυρό λόμπι για την μείωση του ενδιαφέροντος για τα τρόφιμα και την μαζική εισαγωγή τροφίμων από τρίτες χώρες, γιατί πολλοί καρπώνονται τα ωφέλη τέτοιου εμπορίου. Είδαμε τι συνέβη με την μεταρρύθμιση αγορά ζάχαρης. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποκύψει και να ενδώσει στις πιέσει αυτού του λόμπι. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει υπόψη την ασφάλεια των τροφίμων και τη πολιτική ε, τροφίμων, γιατί μερικές φορές τα λόμπι ε, δεν ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά μόνο για τα προσωπικά τους ε, συμφέροντα και κέρδη. Ε, Κύριε Πρόεδρε, το εμπόριο κανονικά θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και του δίκαιου. Και αυτό θα ήταν πολύ καλός λόγος ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε τις πολιτικές για να περιορίσουμε και την ένδια και τις επιστημιστικές κρίσεις. Η Γεωργία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα νέα κράτη-μέλη ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι άμεσες πληρωμές για τις χώρες αυτές είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι για τις παλιές χώρες. Και ερχόμαστε να ανταγωνιστούμε τους παραγωγούς Λατινικής Αμερικής που δεν έχουν τα ίδια ποιοτικά πρότυπα και ε, έχουν και χαμηλούς στασμούς. Η δική μας ανταγωνιστικότητα λοιπόν πλήττεται, γι' αυτό και υποστηρίζω την έκθεση γιατί ζητά αναθεώρηση των εμπορικών πολιτικών και παρακολούθηση, έλεγχο, ίδιες προδιαγραφές για τις ε, τρίτες χώρες με εκείνες τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόνο τότε να ανοίγουμε τις αγορές μας για τα προϊόντα τους, εφόσον έχουμε αντιστάθμιση των αποζημιώσεων από τις αγωγές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν μιλώ με πολλούς φίλους που έχω στις φτωχές χώρες του κόσμου, λέω τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε να ακουφίσετε τη φτώχεια στη χώρα σας. Πολύ συχνά μου λένε, όχι αναπτυξιακή βοήθεια, αυτό που θέλουμε είναι να βοηθήσετε τους επιχειρηματίες στη χώρα μας να δημιουργήσουν πλούτο εδώ και να μπορούν να συναλλάσσονται εμπορικά με την Ένωση, να ανοίξετε τις αγορές σας. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα εδώ είναι ότι έχουμε την κοινή γεωργική πολιτική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα σωρό επιδοτήσει και εκείνοι. Αλλά ε, είμαστε υποκριτέ, κρίνουμε τι αγορέ μα στην πάρα πολύ καλή παραγωγή από αναπτυσσόμενε χώρε. Και επίση βάζουμε και προδιαγραφέ που τι λέμε υγιεινεί και φυτογειονομικέ. Μα πολύ συχνά το χρησιμοποιούν αυτό ως εμπόδιο μη δασμολογικό απέναντι στις αγωγές από τρίτες χώρες, αναπτυσσόμενες. Είναι ε, καιρό να εμπιστευτούμε τους καταναλωτές. Ας επιλέγουν οι καταναλωτές τι θέλουν να καλλιεργούμε στην Ευρώπη αλλού και ας σταματήσουμε τις επιδοτήσει ζημιογόνων ε, καταστάσεων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μοναδική στο ότι έχει γραφειοκρατία, ε, διαφθορά, υποκριτία, ε, αμυθικότητα μάλιστα. Στο τέλος της δεκαετίας του 50 ο πρέσβης Αργεντινής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο εκπρόσωπος των αντιζωμένων χωρών και είπε τότε ότι αν θέλετε να επιδοτείτε τους γεωργούς σας το κατανοούμε αυτό. Ε, μπορεί να μας αρέσει αλλά το κατανοούμε, αλλά παράλληλα όμως μη μας δίνετε και διπλό ράπισμα με το να φέρνετε τα δικά σας τα πλονάσματα στις δικές μα αγορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το άκουσε τότε και δεν το ακούει και σήμερα. Ε, Βεβαίω ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να προσφέρει γεωργικά, όπλα, ε, γεωργικά προϊόντα ε, προσφέρει τα όπλα και εξακολουθεί να έχει αυτόν τον προστατευτισμό η κοινή πολιτική υπάρχει από τη δεκαετία του 60 και αυτό το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η οικολογική καταστροφή, η φτώχεια, οι υψηλέ τιμέ των τροφίμων. Ε, τι μπορούμε, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά όταν δίνουμε ε, στους ίδιους οργανισμούς τις ίδιες εξουσίες. Σας ευχαριστώ πολύ κανονικά ε, συμφωνώ 100% ε, και είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα όλα αυτά που είπε ο κύριος Κεμάλ αλλά ε, σήμερα όμως θα διαφωνήσω. Κατέληξα στο ότι η επισητιστική ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, ανάπτυξης του πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ασφαλής ε, στην δική της την ψηφιστική ασφάλεια. Και αυτό σημαίνει αυτάρκεια. Αυτάρκεια όχι απαραίτητα στην παραγωγή αλλά υποπαραγωγή όπου παίρνουμε ε, την τροφή από το στόμα των πεινασμένων. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε την αυτάρκεια στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν λοιπόν έχουμε αυτάρκεια ως στόχο του προγραμματός μας, δεν νομίζω ότι όλα τα άλλα προστίθενται στο διεθνές εμπόριο. Ε, τα τρόφιμα είναι κάτι ιδιαίτερα που δεν, με το οποίο δεν μπορούμε να παίξουμε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση Hostlink ε, Το, ε, οι πρωτενε είναι απαραίτητε. Ε, η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να δραστηριοποιηθεί και να έχει τη δική της παραγωγή πρωτεϊνών. Πρέπει να σκεφτούμε όλε τις δυνατότητε που υπάρχουν από την έρευνα και την καινοτομία, καινοτόμε πρόπτικες μέχρι και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Δεν πρέπει λοιπόν να χάνουμε την, ε, τον κύκλο της οικονομίας. Η Κομισιόν ε, θα πρέπει ε, να άρει την απαγόρευση της χορήγης πρωτεϊνών σε ζωοτροφές. Η επεξεργασία των τροφών αυτών ε, θα πρέπει να υπηρετεί την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή καταστρέφονται πάρα πολλέ πηγέ πρωτεϊνών, απλά και μόνο γιατί δεν είμαστε σε θέση να οργανώσουμε τη σωστή μεταχείριση αυτών των ε, ουσιών. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που εξαιτία της των κακών ε, τροπολογιών που κατατέθηκαν στην καλή έκθεση του κυρίου Χάουσλινγκ τελικά α, ε, χρειάστηκε να την καταψηφίσω και μάλιστα ο ίδιος ο εισηγητής απέσυρε την υπογραφή του από την έκθεση. Λυπάμαι που με τις τροπολογίες αλλοιώθηκε τόσο η έκθεση και έτσι ε, διευκολύνθηκε και η εισαγωγή των γενετικώς τροποποιημένων ε, σπόρων και καλλιεργιών. Δεν θα πρέπει να ενδώσουμε σε αυτή την πίεση γιατί τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα θα είναι απειλή στην δημόσια υγεία. Και συμφωνώ με τον ε, συντάκτη, γι' αυτό και εγώ έκανα ότι και εκείνος καταψήφισε την έκθεση. Ευχαριστώ. Πρώτα ο κύριος Ντεάντζελης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για την έκθεσή της. Το να μιλά κανείς για την ισότητα των δύο φίλων σήμερα στον κόσμο της εργασίας ε, δεν είναι μόνο κάτι το ρηματικό, το ρητορικό. Ε, η απασχόληση των γυναικών στην Ευρώπη είναι θέμα στρατηγικής ε, σημασίας και σε πολιτιστικό και σε οικονομικό επίπεδο εάν ε, βλέπουμε το επίπεδο απασχόλησης ε, των γυναικών, αν ήταν ε, το ίδιο με αυτό των ανδρών, τότε θα αυξάνει το κατά 30% το ΑΕΠ. Η κρίση λοιπόν δεν πρέπει να ανασχετίζει τις προσπάθειές μας, τουναντίον θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ενεργό πολιτική στον τομέα της γυναικείας απασχόλησης. Πολιτικές λοιπόν απασχόλησης που στοχεύουν στο να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις πάνω στην απασχόληση των γυναικών και να προλαμβάνονται κυκλικές αντιδράσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο της πολιτικής ε, για τις ε, γυναίκες. Θα πρέπει να προάγουμε την ε, εκπαίδευση και απασχόληση των γυναικών. Και υπάρχει και άλλο ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, το θέμα της βίας που ασκείται εναντί των γυναικών. Σήμερα η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει μια δική της πολιτική για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις μορφές της βίας εις βάρος των γυναικών. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Tak, Når man Ευχαριστώ. Άκουσα όλη αυτή τη συζήτηση για τις ποσοστώσεις ε, ε, σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείε. Ε, γίνεται πόλεμος χαρακομμάτων αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα. Εγώ ε, κανονικά είμαι κατά των ε, υποχρεωτικών ποσοστώσεων διανόμου γιατί είναι ε, κακό αυτό και για τις εταιρείε, αλλά και για τις αξιόλογες γυναίκες με προσόντα και ικανότητες που περιθεροποιούνται στην ηγεσία τέτοιων εταιριών. Θα μπορούσε κανείς να επιλέξει τη ρεαλιστική άποψη που λέει ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στις εταιρείε πολιτική ισότητας, αλλά να έχουμε δικούς μας στόχους. ή να πούμε κάθε επιχείρηση να ορίζει εκείνη το στόχο της. Αυτό θα είναι καλό και για τις γυναίκες και για τις επιχειρήσεις γιατί ε, θα διαχειρίζονται μόνοι τους στόχους. Ευχαριστώ. Κυρία Σερακιάνη, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα την έκθεση για την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα και, ανάμεσα στη, και για τη γυναική αυτόχεια στην Ευρώπη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα συζητήσαμε σήμερα όλα αυτά ε, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την ημέρα της γυναίκας. Ε, ε, παρά την οδηγία που αφορά στην ισότητα μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία, στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση, υπολείπονται πάρα πολλά για να μπορέσουμε με να επιτύχουμε το στόχο μας. Ε, Παραδείγματος χάρη, το επίπεδο της εκπαίδευσης ε, των γυναικών ε, έχει βελτιωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια και σήμερα ο αριθμός ε, των πτυχιούχων γυναικών είναι πολύ μεγαλύτερος. Όμως παρόλα αυτά οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια απασχόληση όπως και οι άνδρες στις θέσεις απασχόλησης. Είναι αρμόδιες, υπεύθυνε για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους και αυτό εμποδίζουν τις γυναίκες να εργαστούν. Θα ήθελα να κλείσω αναφέροντας ότι θα πρέπει να εκφραστούμε υπέρ, ε, της, ε, υπέρ των γυναικών, υπέρ των ε, οργανώσεων των γυναικών που κατεβαίνουν σήμερα για να διαδηλώσουν. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε να κάνω μια επεξήγηση γιατί καταψήφισα το ψήφισμα αυτό που κάνει μια αξιολόγηση του 2010 υπό τη σκοπιά της ισότητας. Φυσικά είμαστε υπέρ της ισότητας ανδρών και γυναικών, αλλά το είστε υπέρ και της άμβλωσης, της ε, επιλογής, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, που λένε ότι η άμβλωση ουδέποτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως τρόπος ε, ε, ρύθμισης της γεννητικότητας η υιοθέτηση ενό τέτοιου ψηφίσματος ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταστρατηγεί τι ε, αρμοδιότητε των κρατών μελών και ε, προδικάζει και το δικαίωμα επιλογής στη ζωή. Λυπάμαι που η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υποστήριξε το κείμενο. Είναι πολύ ανησυχητικό μήνυμα και έγινε μια πρόταση από οργανώσει προ του ευρωβουλευτέ που εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα επιλογή να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση αυτή. Ο κύριο Στάκουλα. Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το θέμα τη ισότητα των ανθρώπων και γυναικών, όχι μόνο σήμερα στον εορτασμό τη Παγκόσμια ημέρα τη γυναίκα. Το θέμα αυτό θα πρέπει να μα απασχολεί μόνιμα. Επίσης ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαφορά μεταξύ των ανδρών και των γυναικών είναι παράγοντες που ε, μας εμπλουτίζει, αλλά οι άνδρες είναι ίσοι με τις γυναίκες. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε αυτό το θέμα της ισότητας και θα πρέπει αυτή η ισότητα να χαρακτηρίζει όλε τι πτυχέ τη ζωή μα. Θα πρέπει και στην αγορά εργασία οι άνδρες ε, και οι γυναίκε να την χάνουν ίση μεταχείριση. Μέχρι στιγμή, ε, δυστυχώ η κατάσταση έφερε τι γυναίκε σε μια ασθενέστερη κατάσταση και ω προ του μισθού και ω προ άλλου παράγοντε. Δεν θα πρέπει οι γυναίκε να είναι το ασθενέ φύλλο. Θα πρέπει να αναγνωριστεί η ισότητα. Και ω προ τι ποσοστώσει. Χρειαζόμαστε ποσοστώσει από τη στιγμή που δεν έχουμε πραγματώσει την ισότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα εγκρίναμε άλλη μια πρωτοβουλία. Ε, αλλά όπω είπε και η Επίτροπος θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Παρά τα μέτρα παραμένει η ανισότητα. Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες είναι πιο μορφωμένες με καλύτερα αποτελέσματα σύμφωνα με τα στοιχεία των πανεπιστημίων. Αλλά συνεχίζουμε να είμαστε να εφιστάμεθα διακρίσει και οι μετανάστριες υφίστανται διπλή διάκριση και μάλιστα σε μεγάλη ηλικία. Ε, ε, σήμερα ακούσαμε πολλές διακηρύξεις, πολλές δηλώσεις, αλλά δεν δίνουμε το παράδειγμα. Αρκεί να αναλύσουμε το ε, φίλο του Προέδρου ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις Προεδρίες, το μόνιμο Πρόεδρο, την Προεδρία του Κοινοβουλίου, του Ελεκτικού Συνεδρίου, τους Επιτρόπους, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει καμία γυναίκα. Ή οι Προεδρίες ε, εδώ των πολιτικών ομάδων ή η απουσία γυναικών στις αντιπροσωπείες κάποιων χωρών. Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να είναι ανδρική. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο, γι' αυτό υποστήριξα αυτή την προσπάθεια και πιστεύω στις αντιπροσωπιες καποιων χωρων η εικονα της ευρωπαικης ενωσης συνεχιζει να ειναι ανδρικη θα πρεπει να προχωρησουμε πολυ περισσοτερο γι αυτο υποστηριξα αυτη την προσπαθεια και πιστευω στις ποσοστωσεις σε αυτό το δύσκολο δρόμο ιδιαίτερα, όπως είπαμε, τα λόγια στα έργα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βαϊντέρα, για ένα λεπτό. Lai gan stāvoklis sieviešu tiesību jomā ir uzlabojies, tomēr vēlos no... Η κατάσταση σε θέματα γυναικών έχει βελτιωθεί και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τρία πράγματα που πρέπει να εξετάσουμε. Το ένα είναι η αμοιβή τους, η αποζημίωσή τους. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Οι διαφορές αυτές επιτάθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης γιατί υποστηρίξαμε τις τράπεζες αλλά όχι τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Δεύτερον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το ποσοστό ε, γονιμότητας ε, είναι πάρα πολύ χαμηλό, δεν υπάρχει υποστήριξη των γυναικών και τρίτον στην ε, απασχόληση ε, το, ο ιδανικός λόγος θα ήταν 50-50 αλλά υπάρχουν πολύ λίγες γυναίκες. Όλα αυτά τα βλέπουμε και στις ηγετικές θέσει σε πάρα πολλούς οργανισμούς. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή δεν προχωράει αρκετά. Ευχαριστώ. Εγώ λοιπόν υπερψήφισα την έκθεση και υπερψήφισα και το θέμα των ποσοστώσεων. Και θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω την κυρία Ρέντινγκ ε, για το ότι απαιτεί να ληφθούν ε, μέτρα και σε επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να εφαρμοστεί Εκεί λοιπόν έτσι καλώς προβλέπεται η ισότητα των δύο φύλων. Θεωρώ ότι στη δημοκρατία δεν πρέπει να είναι απαραίτητε οι ποσοστώσει, όμω αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Ήδη πριν από 10-15 χρόνια εισήχθησαν σε εμά οι ποσοστώσει, τότε διαφωνούσαμε, αλλά εντωμεταξύ διαπιστώσαμε ότι οι ποσοστώσει βοηθούν στο να λειτουργεί ε, η κατάσταση υπέρ των γυναικών. Οι γυναίκε βρήκαν θέσει απασχόληση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που ήρθατε και αντικαταστήσετε την Αντιπρόεδρο και ευχαριστούμε και τους διερμηνείς. Η πρόσφατη απόφαση που λέει ότι απαγορεύεται διακριτική μεταχείριση ε, για θέματα φύλου και άλλες αιτίε. έχει τόσα ελαττώματα σε πολλά επίπεδα και δεν ξέρουμε πού να αρχίσουμε. Καταρχήν, ως προς το κόστος, θα αυξηθεί και το κόστος και των ασφαλίστρων. τι γίνεται σχέση με την ομολογία του 10 ως προς την ομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και μάλιστα με τις οδηγίες ε, υπέρ της διακριτικής μεταχείρισης και εκεί υπήρχε πρόβλημα με το αναλογιστικό σύστημα. Φαίνεται ότι έγινε σύγχυση μεταξύ του γράμματος και του πνεύματος του, του νόμου. Βέβαια, δεν θα πρέπει το κράτος ε, να ε, μπαίνει στη μέση και να χαρακτηρίζει τι συναλλαγέ παράνομε. Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη τελική ανάλυση. Κάθε χώρα μπορεί να έχει του δικού κανόνε ε, για την ισότητα των φύλων ανάλογα με τι δικέ δημοκρατικέ ε, διαδικασίε. Γιατί ένα ανώτατο δικαστήριο μερικέ φορέ μπορεί να γίνει τυραννία όταν προσπαθεί να τα ελέγξει όλα. Eh, Κύριε Πρόεδρε, η ε, γυναικεία φτώχεια είναι μια κατάσταση που ανάγεται στο παρελθόν και σίγουρα δεν είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Εγώ λοιπόν υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου Πλάμπ γιατί είμαι πεπισμένος ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο ισχυρή δέσμευση για να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος προς την κατεύθυνση της ισότητας των δύο φύλων. Πιστεύω ότι τα μέτρα που ελαμβάνονται σε αυτή την έκθεση θα συμβάλλουν σημαντικά ίσως όχι καθοριστικά, αλλά ένα βήμα προς τα μπρος, ε, προς την κατεύθυνση μιας Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισότητα των Δύο Φύλων. Η τα κράτη-μέλη ε, έχουν και πρέπει να προάγουν συγκεκριμένα προγράμματα ε, που αφορούν ε, στην συμπερίληψη των γυναικών στην αγορά εργασίας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Είναι καθοριστική σημασία στα προγράμματα αυτά να συντονίζονται όχι μόνο σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο αλλά να υπάρχει συντονισμός και με εξωτερικούς εταίρους πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η γυναίκα ανέκαθεν έκανε την αόρατη δουλειά ε, στο σπίτι ε, και επίσης φροντίζει αυτά που δεν μπορούν ούτε να αγοραστούν ούτε να μετρηθούν τα άειλα, τις άειλες αξίες. Ε, Παρ' όλα αυτά παραμένουμε με ε, φτώχεια και με κίνδυνο φτώχεια που πλήττει ιδιαίτερα στην οικονομική κρίση τις γυναίκες. Ε, οφείλουμε να ε, εκριζώσουμε τη φτώχεια των γυναικών. Γι' αυτό υποστήριξα την πρωτοβουλία με εκείνα τα μέτρα και τις νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες που απαιτούνται. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές ενεργητικές των γυναικών με κοινωνική προστασία και με ειδική προσοχή στις πιο ηλικιωμένες και ε, στις γυναίκες με αναπηρία. Να συμμετέχουν ε, να ευνοήσουμε τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας γιατί είναι ε, προς όφελος Και θα αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 13% όπως το δείχνουν διάφορες μελέτες αν γίνει αυτό. Είναι θέμα δικαιοσύνης αλλά κυρίως είναι μια ευκαιρία για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφοι. Η συνεδρία διακόπτεται ως τις 3. Καλό μεσημέρι. Thank